Καλησπέρα. Γιατί πολύ μεγάλο έχει Λοιπόν, θα ψηφίσουμε αμέσως την έκθεση Μιγκόλσκι. «17 Σεπτεμβρίου είχε υποβληθεί 345 τροπολογίες αρχικά και με τους σκιώδεις προσπάθησε ο εισηγητής να δημιουργήσει συμβιβασμό, να αναλάβει όσο δυνατόν περισσότερες, 18 συμβιβαστικές που όμως δεν τις δέχονται όλοι. Δεν τις δέχονται. Λοιπόν θα είναι δύσκολη ψηφοφορία και γι' αυτό παρακαλώ βγάλτε ήδη τις κάρτες σας Λοιπόν, στην αρχή η έκθεση Μιγκάλσκι αναφερόταν σε πολλά προηγούμενα και παραδείγματα και τελικά είπαμε να μην γίνει έτσι μια υπερφορτωμένη έκθεση, να συμπυκνωθεί κάπως Τη συμπίκνωσε ο κύριος Μιγκάλσκι, αλλά κατατέθηκαν 345 τροπολογίες και πολλές από αυτές τις καλύπτουν οι συμβιβαστικές βέβαια. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Μικάλσκι οι συντάκτες των τροπολογιών ανέμεναν να συμπεριληφθούν όλες τις συμβιβαστικές, αλλά δεν γινόταν βέβαια αυτό. Για να είναι η έκθεση πιο εύληπτη, χρειάστηκε η συμπίκνωση, δεν φταίει ο κύριος Μιγκάλσκι. Οπότε παραλαμβάνω, οι συνάδελφοι που λένε ότι η έκθεση δεν είναι πια τόσο αναγνώσιμη, έχει πολύ περισσότερα ή αντιφατικά στοιχεία, παρακαλώ να καταλάβουν ότι είναι δική τους ευθύνη, γιατί αυτοί το προκάλεσαν διότι υπέβαλαν τροπολογίες οι οποίες εν μέρη ελήφθησαν υπόψη από τον κύριο Μιγκάλσκι για να μην υπάρξει ανησυχία και αντιρρήσεις. Ε, θέλω να το πω αυτό γιατί ακούω κάποιες φήμες να κυκλοφορούν. Λοιπόν, να κάνω μια έκκληση ούτω ώστε όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία να λάβουν υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύνολο. Ε, ή καλύτερα έχει γίνει πιο ευρεία και έχει γίνει πολύ πιο εκτεταμένη σε σχέση με το παρελθόν και ιδιαίτερα τότε ε, και ιδίως από τότε που μπήκαν οι ε, χώρες μέλη της Ανατολικής Ευρώπης που οπωσδήποτε είχαν υποστεί πολύ χειρότερα από 50 χρόνια και βεβαίως επειδή έχουν γίνει πολλές τροπολογίες μπορεί να είναι λίγο δυσνόητη η έκθεση. Το καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ να σκεφτείτε πώς θα συμπεριφερθείτε ο καθένας από εσάς. Σας παρακαλώ. Εγώ πιστεύω δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε να αποκλίνουμε αλλά να βοηθήσουμε αυτούς που έκαναν την προσπάθεια να αναγνωρίσουμε την προσπάθειά τους και να αναγνωρίσουμε ότι οι συζητήσεις με τους Κιώδης ήταν πολύ έντονες και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αφαιρέσουν οποιοδήποτε λόγο να είναι κανείς κατά της έκθεσης. Με συγχωρείτε που τα ανέφερα αυτά τόσο αναλυτικά, αλλά ήθελα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να καταλάβετε τι ακριβώς θα γίνει τα επόμενα λεφτά. λεπτά. Ο κύριος Μιγκάλσκι θα ήθελε να προσθέσει τίποτα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να σε ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτά που μόλις είπατε. Πραγματικά έχω την εντύπωση ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πετύχουμε συμβιβασμό. Τελικά, ο συμβιβασμός δεν μπόρεσαμε να, τον, να μπόρεσε να επιτευχθεί σε όλα τα σημεία της εκθέσεως. Οι διαφορές μεταξύ κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης από τη μία με τη δυτική Ευρώπη είναι διαφορές που εξακολουθούν να εφίστανται. Οι συμβιβασμοί μου σχεδιάστηκαν ούτω ώστε να γεφυρώσουν αυτές τις διαφορές. Καμιά φορά όμως οι προσπάθειές μου ήταν μάταιες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους προσπάθησαν να συμφωνήσουν και να έχουμε μια κοινή έκθεση και μόνο η ψηφοφορία τελικά θα δείξει πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν. Ευχαριστώ. Να κάνουμε συζήτηση τώρα από αυτού. Πολύ σύντομο σχόλιο κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να υπονομεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μενέντεθ, σκιώδης των σοσιαλιστών, αντιμετώπισε αυτό το δύσκολο κείμενο πολλές από τις συμβαστικές προτάσεις που απέστειλε στον κύριο και τις έστειλε θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να απορριφθούν. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν τη συμβολή του κυρίου Μενέντεθ στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο. Α, το ανέφερα και σήμερα το πρωί στην κυρία Κάμεβατ. Ορίστε. Κοιτάξτε, αν ε, τόσο γρήγορα θέλατε πάντα να κάνουμε ψηφοφορίες όπω τώρα, εν πάση περιπτώσει υπενθυμίζω ότι η γραμματεία τη Επιτροπή είπε ότι στο κατάλογο ψηφοφοριών κάτι ξεχάσαμε. Μετά την τροπολογία 29 Σάντσε Σμιθ πρέπει να προσθεθεί 28 του κυρίου Καβαντά. Ε, Έπρεπε να το αναφέρω κύριε Καβαντά. Θα ψηφίσουμε και τη δική σας τροπολογία λοιπόν. Οπότε, λοιπόν, Ξαναλέω, αν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Λοιπόν, ε, ένας ΕΛΚ είναι παραπάνω. Εντάξει, εξής, μάλιστα, να μην ψηφίσετε, μάλιστα. Εντάξει, ο Μάταλα μπορεί να ψηφίσει, ωραία. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία. τέσσερα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Δώδεκα δεκατέσσερα απορρίπτεται. Κοιτάξτε, ψηφίζουμε. Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ποιο δεν ψηφίζει. Λοιπόν, 12-14, αλλά δεν δούλευε το μηχάνημά σα. Είστε υπέρ κατά. Σε παρακαλώ προσπαθήστε. Να ελέγξουμε γιατί υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Υπέρ παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται. 178. Υπέρ. Κατά. Ίδιος συσχετισμός απορρίπτεται. Κυρία Κουλάμ, δεν έχετε την κάρτα σας. Α, μάλιστα. Α, ωραία. Αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ωραία. 180 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται 176 άρχεται ο έλεγχος της 176 υπέρας. 13 υπέρ 13 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. 13-11 δηλαδή, μάλιστα. Μάλιστα γιατί δουλεύει ένα μηχάνημα. Ωραία. Λοιπόν και πάλι. Τι γίνεται. Μα δεν δουλεύει το μηχάνημά σα. Δεν δούλεψε. Καλά. Ξαναρχίζουμε. Και παρακαλώ τους τεχνικούς να μας βοηθήσουν. Άρχεται η ψηφοφορία 176. Πέρας. 13 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται. Ωραία, 13 υπέρ, 15 κατά μέσα 182 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος, άρχεται. 182. Πέρας. 11 υπέρ, 17 κατά, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά τι και πάλι συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η 188 ελέγχεται πέρας απορρίπτεται 12 υπέρ 17 κατά 100 Λοιπόν, περνάμε στη 200. Υπέρ είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται για τη 200. Πέρας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε όταν πρέπει. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 15-14 εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται για τη 206 πέρας 11-18 απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές έλεγχος α απορρίπτεται συγγνώμη 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 216 πέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολόγηση της 211. Ορίστε, παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω μετά τα διδακτικά προγράμματα τη φράση τονίζει ταυτόχρονα ότι η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση θα, στην ίδια προσέγγιση θα πρέπει να κινηθούν για, ε, όσον αφορά την, ε, την κρίση των διαφόρων καθεστώτων του κομμουνισμού και του σελισμού στην τελευταία σελίδα να γίνει αυτή η προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 212. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ. όχι. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 και υπόλοιπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 232 κάτω Εμίλιο Μέντες βάλει υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για μια ακόμη φορά 15 συμβιβαστική 15 Ψηφ, ψηφοφορία πέρας 16-12 απορρίπτεται όπως είχα προβλέψει. 234 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας 17-12 εγκρίνεται στην άλλη σελίδα 247 247 Καβαδά Σμιθ υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 247 πέρας 13 ψήφοι με 11 εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 248 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 13 με 11 εγκρίνεται. 249 επέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 249. Πέρας. 13-11 εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200 50 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 250 έρχεται πέρας 13 με 15 απορρίπτεται 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 ναι 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ τι θέλετε εγκρίθηκε εγκρίθηκε με τη συμβαστική 16 ξεχάστε την εντάξει ωραία 256 υπέρ κατά να με βοηθάτε γιατί αλλιώς χάνομαι. 251 υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος γιατί 251 έρχεται. Πέρας. 14-12 απορρίπτεται, 261 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 200, έλεγχος, 261, άρχεται η ψηφοφορία για τη 261 πέρας 12 με 15 απορρίπτεται το είπα το είπα 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή μάλλον ξεκινάμε έλεγχο πέρας 10 με 16 απορρίπτεται 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 264 άρχεται ψηφοφορία πέρας 15-10 εγκρίνεται 265 και υπόλοιπε μέχρι τη 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 287 ελέγχουμε τη 286. Άρχεται η ψηφοφορία τη 286. Πέρας. 15 με 14. Ε, συμβαίνουν αυτά. Ωραία, εγκρίνεται. 287 υπέρ. Α 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 297 υπέρ 296 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας είναι σαφέστατο το αποτέλεσμα 22 με 7 αγαπητέ 297 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 298 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 299 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 18 πέρας 13 με 16 απορρίπτεται πάμε στην 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος μάλλον για 301 άρχεται Ψηφοφορία πέρας. 15 με 14 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Μάλιστα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την συμβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 με 13 εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 319 άρχεται. πέρασε. 19 με 7 εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 332 υπέρ κατά όχι. Συμβιβαστική 20. Α, το πήγα πολύ γρήγορα. 22. 22. Όχι 22. Συμβιβαστική 20. Μα πού είναι αυτή το πράγμα. Α, ναι, 20, 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 332 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση έλεξε 14-15 απορρίπτεται 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 337 όχι 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 334 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 16 με 13 εγκρίνεται 335 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται επαλήθευση μάλλον. 16-13 εγκρίνεται. 338 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 348 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 351 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Για την 351. Έληξε. 12-16 απορρίπτεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 354 υπέρ κατά χες επαλήθευση 12 με 17 απορρίπτεται 355 υπέρ κατά χες επαλήθευση 12 με 16 απορρίπτεται. 21 υπέρ. Όχι. Α, όχι 17. 17, ε. Ούτε. Δεκατέσσερα, δεκατέσσερα υπέρ, κατά, επαλήθευση. 15 με 14 εγκρίνεται 24 α όχι 25 25 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται παλήθευση καλά παλήθευση της 20 της 26. 15 με 14 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά yes. 14 με 12 εγκρίνεται. «28 υπέρ κατά προχές εγκρίνεται». «30 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται». «31 υπέρ κατά προχές επαλήθευση». 17 με 10 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά χες επαλήθευση. 15 με 14 εγκρίνεται. Τώρα 47 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αρχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αρχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αρχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αρχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αρχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Δεκατέσσερις με 13 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά χες επαλήθευση. 15 με 13 εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, επαλήθευση. 15 με 13 εγκρίνεται. 73 υπέρ. Αφού μόλις κάναμε την 69 Α, ναι, ναι. Α, μάλιστα ναι. Πιο δύσκολα τώρα. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ όχι 85 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 85. 10 με 19 απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά οχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 91 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά οχές απορρίπτεται επαλήθευση μάλλον 13 με 14 εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απαλήθευση Δεκαπέντε με 14 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά ποιες επαλήθευση. Για τη συμβιβαστική 7 12 με 17 απορρίπτεται. 116, 17, 18, 19 υπέρ, κατά, ποιες επαλήθευση. 14 με 15 απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Α, όχι, όχι, όχι, Α, ναι, ναι, ναι. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ε, επαλήθωση. 12 με 17 απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση. 10 με 19 απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται. 125 υπέρ τα χες επαλήθευση. Πέρας 18 με 11 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για τη συμβαστική 8. Πέρας 16 με 13 εγκρίνεται. 120, 139 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. 11-18 απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος άρχεται. Πέρας. 16-13 εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε άρχεται για τη συμβαστική 10 έλεγχος. Πέρας. 14-15 απορρίπτεται. 151 και 152 υπέρ. Κατά. Έλεγχος άρχεται. Πέρας. 14-15 απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται. Πέρας 15-13 εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται πέρας 12-17 απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. 13-16 απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 5 με 24, με συγχωρείτε, ήταν σαφής ο συσχετισμός. 169 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 13-16 απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται για την 173 πέρας 13-15 απορρίπτεται 1 και 2 1 και 2 υπέρ κατά Ένα και δύο και πάλι παρακαλώ υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Έλεγχος της πέντε. Πέρας. 12-17 απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές ε, ναι, εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Πέρασε. 9 προς 19. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται για τη 10. Πέρας. 13 προς 14 απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά ε, μα δεν δε βλέπουμε. Ε, λοιπόν, ψηφίζουμε την 11. Πέρασε. 12 προς 14 απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος άρχεται. Πέρας. 13-14 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος άρχεται. 10 10-18. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Άρχεται. 11 προ 13. Απορρίπτεται. Ψηφίζω κατά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει η πρόεδρος. Άλλη μία ψήφος κατά. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου, ψήφισα κατά. Καλά, δεν πειράζει. Κύριε Μιγκάλσκι. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω απόσχει στην τελική αυτή ψηφοφορία. Απήχα στην τελική ψηφοφορία διότι δεν μπορούσα να υπερψηφίσω μία έκθεση το περιεχόμενο της οποίας δεν ήταν αληθές. Εκπλήσωμαι και ανησυχώ για τρία πράγματα. Που τα πράγματα αυτά σχετίζονται με την εξίσωση του κομμουνισμού με τον ναζισμό αντί να γίνεται μία αναφορά σε στρατόπεδα θανάτου των ναζί έγινε απλώς μία αναφορά σε στρατόπεδα θανάτου και η έλλειψη αναφοράς, υπήρξε και έλλειψη της αναφοράς της φαγής του Κατίν. Ευχαριστώ εκείνους οι οποίοι υπερψήφισαν, αλλά αυτή η έκθεση δεν πρόκειται να έχει την υπογραφή μου, διότι θα ήταν κάτι για το οποίο θα αντρεπόμουν. Ο κύριος Καβαντά. Πολύ σύντομα. Πριν την ψηφοφορία εφιστήσατε την προσοχή μας σε ένα ενδεχόμενο ότι δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι δεν ε, γνωρίζουν αρκετά την ιστορία της κεντρικής Ευρώπης. Διαφωνώ. Αν ήταν ε, επιθυμία θα συμφωνούσα, αλλά είναι διαπίστωση, διαφωνώ, ε, πολύ γνωρίζουμε και εγώ ο ίδιος που έχω εργαστεί πολύ σε αυτές τις χώρες και δεν θέλω με κανένα τρόπο η πολιτική να γράφει την ιστορία. Γιατί είδαμε που καταλήγουμε και μετά την ψηφοφορία θα πρέπει να πω στον κύριο Μιγκάλσκι ότι δεν είναι ότι παραγνωρίζουμε την ιστορία που ήταν δραματική αλλά δεν πρέπει να ξαναβάζουμε το ατσάλι στη φωτιά. Εάν η έκθεση αυτή αφορούσε μόνο την ιστορία της εκπαίδευσης των νέων θα είχε υπερψηφιστεί από όλε τις ε, πλευρές του σώματος. Εάν θέλει να καταδικάσει ιστορικούς, κάποιες ελίτ, κάποιου διανοούμενου, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι αυτό που κάναμε δεν είναι επειδή θέλουμε διχασμό, αλλά είναι θέμα αλληλεγγύη με τα μαρτύρια των λαών της ε, Κεντρικής Ευρώπης που πλήρωσαν με το αίμα του ε, τα μαρτύρια των λαών τη Δύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόκιος. Yes. Η Πρόεδρο, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και εν γέννη συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μεγκάλσκι ε, πρόκειται και για πιο σημαντικά θέματα, για περισσότερα πράγματα που τίθενται. Δεν θα ήθελα να καταδικάσω κανέναν, όμως πρέπει να διαπιστώσω ότι υπάρχει κάποια σχιζοφρένεια εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ή αυτό, ή αγνοεί κάποια πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ενήμερο για όσα συμβαίνουν και όσα έχουν συμβεί. Πάμε στην κατάσταση που κρατούσε πριν το 2009. Τι συνέβη το 2009. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα κείμενο σχετικά με τη συνείδηση και τη μνήμη όσον αφορά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ήταν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο ψήφισμα αυτό με στον ίδιο βαθμό αποτιμήσαμε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντιμετωπίσαμε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα με τον ίδιο τρόπο. Το δύο, η προσέγγιση των δύο μέτρων και δύο σταθμών καταργήθηκε χάρη σε αυτή την επανάσταση. Και έχω την εντύπωση ότι μετά το 2009 που ξεκίνησε νέος κύκλος, λοιπόν με τη νέα θητεία, υπαναχωρήσαμε, επιστρέψαμε σε παλιές θέσεις. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. όσον αφορά την ε, αξιολόγηση της ιστορίας και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ανησυχητικό διότι αυτό που παρατηρούμε σήμερα στη Ρουμανία είναι μια υπαναχώρηση, επιστροφή στα παλιά. Μια πλειοψηφία δύο τρίτων ε, υποστηρίζει τον κομμουνισμό. Και πρέπει να φοβόμαστε. Φοβόμαστε ότι οι κομμουνιστικές δυνάμεις και οι μετακομμουνιστικές δυνάμεις ξαναέρθουν στην εξουσία. Και η διαδικασία που ξεκίνησε το 1989 θα σταματήσει ξανά ή θα ε, τεθεί τροχοπέδι σε αυτή τη διαδικασία. Και το λέω αυτό σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου, μία μέρα που γιορτάζουμε την εξέγερση, τη λαϊκή επανάσταση που ξεκίνησε στην Τιμισοάρα τότε και το μήνυμα που στέλνουμε είναι πολύ κακό. Ευχαριστώ τον κύριο Μιγκάλσκι, τους αγαπητού συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν και εύχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δει τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Και η ιστορία της Ευρώπης, στον οίκο τη Ευρώπη, Ευρώπης, της ιστορίας της Ευρώπης, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ιστορία μας. Είτε η ιστορία αφορά την Ανατολική Ευρώπη, είτε αφορά την Δυτική Ευρώπη. Η αφήγηση τη ιστορία πρέπει να είναι παρόμοια. Ευχαριστώ κύριε Τόκιο. Ο κύριο Βάτιμο και μετά ο κύριο Μπορώ να μιλήσω. Είμαι ανάμεσα εκείνους που καταψήφισαν αυτή την έκθεση από την αρχή τη θεωρούσα ένα εγχείρημα ρητορικό άχρηστο. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια επίσημη ιστορία της Ευρώπης. Σε πολλά σημεία, πολλά σημεία της εκθέσεως αναφέρεται η ιδέα ότι πρέπει ε, να είναι αντικειμενική και πραγματική η ιστορία. Ποιος το κρίνει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να απαγορεύσουμε την ελευθεροτυπία του τρόπος αν υπάρχει κάποια ανώτατη αρχή που κρίνει τι είναι σωστό, τι είναι αληθές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πολλά από αυτά τα άρθρα αναφέρεται η ιδέα να δημιουργήσουμε ένα κάποιο δικαστήριο που θα κρίνει τις πράξεις. Σε αυτή την έκθεση πολύ συχνά αναφέρεται ότι πρέπει να καταγγείλουμε τα ολοκληρωτικά καθ... καθεστώτα και τα εγκλήματά τους. Και αυτά που δεν από ολοκληρωτικά καθεστώτα, οι βομβαρισμοί των Αμερικανών στο Ιράκ, ότι η Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία εισέβαλαν στη Λιβύη. Τι θέλω να πω, τι είδους επιχείρηματα είναι αυτά. Ε, από τη στιγμή, δηλαδή από τη στιγμή που είναι ένοχα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε Είπα από το 89 μέχρι το 2009 μέχρι σήμερα άλλαξαν κάποια πράγματα σίγουρα, διότι άλλαξε η κρίση μας που θριαμβολογούσε παλιά για τη δυτική δημοκρατία. Κανείς δεν πιστεύει σε αυτά πια. Οι φτωχοί συνάδελφοι της Ανατολικής Ευρώπης αξίζουν κάθε αλληλεγγύη. Εγώ, αν ήμουν ένας Ούγγρος της εποχής παλιάς, θα ήμουν φιλοαμερικανός πλήρως. Αλλά σήμερα δεν μπορεί πια κανείς να είναι φιλοδυτικός έτσι ε, ανοιχτά όπως νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Το καπιταλιστικό σύστημα ε, μας έκανε να καταστρέφουμε από πείνα, από χρέη που δημιούργησε αυτό το σύστημα. Αρκετά φτάνει. Ας μην συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το μύθο της δυτικής απελευθέρωσης κλπ. Εσείς υποφέρατε πολλά στην Ανατολική Ευρώπη και εγώ ντρέπομαι εσάς. Αλλά και εγώ τι να κάνω. 20 χρόνια φασισμό είχαμε στη χώρα μου. Έτσι είχαν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα αυτό, αυτό που είναι εσφαλμένο στην αρχή ήταν η ιδέα να δημιουργήσουμε μια επίσημη πραγματική ιστορία της Ευρώπης από πλευρά ενός πολιτικού οργάνου. Ο συνάδελφο πριν είπε, δεν θέλω να, την ιστορία την αναλαμβάνει πολιτική ακριβώ. Την ιστορία την αναλαμβάνουν ιστορική ή πανεπιστημιακή εκείνοι που μελετούν και εκείνοι που την έζησαν. Ε, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολιτικοί ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριος Λόκεργαρτ. Θα είμαι σύντομος. Και εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι ότι θέλουμε να τιμήσουμε τα γεγονότα του 89 και ότι δεν υποστηρίζουμε αυτούς που, αυτούς που καταδικάζουν αυτά που συνέβησαν στην Ανατολή. Δεν πρόκειται περί αυτού. Συμφωνώ με τον κύριο Βάτη μου για μια φορά. Αυτά όμως πρέπει να τα αποφασίσουν οι ιστορικοί. Βεβαίως. Θα υποστήριζα μια έκθεση που να καταδικάζει αυτά που έγιναν στην Ανατολή, αν ήταν το μόνο θέμα του οποίου θα ψηφίζαμε. Η έκθεση αυτή δεν εστιάζει επαρκώς. Είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι σαν να στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο με αυτή την έκθεση. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε τέτοιου είδους χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο εστιασμένοι αν θέλουμε να πούμε κάτι πολιτικά για ένα τέτοιο θέμα. Και γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση, γιατί όπως είπε και ο κύριος Καβαντά και ο κύριος Βάτιμο, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, να καταδικάσουμε τα πάντα αν έτσι επιλέξουμε να δράσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ρόλος μας ως Κοινοβουλίου. Πρέπει να είμαστε σαφείς τι ψηφίζουμε. Αν θέλαμε να ψηφίσουμε για κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα και περιορισμένα αυτά που θα λέγαμε. Ευχαριστώ. Η τελευταία ομιλήτρια η... είναι η κυρία Νεβεντάλογα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η συζήτηση, την έχουμε κάνει τρεις φορές. Όλοι γνώριζαν ότι η ψηφοφορία θα ήταν όπως ήταν. Ο κύριος Μεγκάλσκι, τον κύριο Μεγκάλσκι του οφείλουμε σεβασμό, κάναμε όλοι ό,τι μπορούσαμε και εκείνος, αλλά ξέραμε από πριν τι θα γινόταν. Νομίζω ότι έγινε σοβαρή συζήτηση που δεν χρειάζεται να την απαγορεύουμε τώρα. Ο Χάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Όταν μπήκαμε στο θέμα της έκθεσης αυτής, το ξέραμε ότι θα έχουμε προβλήματα και προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Ήμουν εισηγητής δύο φορές όσον αφορά αυτά τα επίμαχα ζητήματα. Οι διάφοροι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για την ε, ιστορία της Ευρώπης. Εγώ είμαι Φιλανδός και στη χώρα μου ε, υπάρχει κατανόηση για τη θέση του κ. Μιγκάλσκι. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί του, όμως ε, κατανοώ αρκετά τις απόψεις του. Σε άλλα μέρη της Ευρώπης είναι διαφορετική η πραγματικότητα. Ακόμα και ιστορικοί παλεύουν και προσπαθούν να βρουν μία και μοναδική αλήθεια. Όμως γνωρίζω αρκετά για την ιστορία της Πολωνίας, ούτως ώστε να ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές. Πιστεύω ότι η ελευθερία της συνείδησης, η ελευθερία της άποψης σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει για τον κομμουνισμό. Φοβούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε οι μεν τους διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο, διαφορετικές νοτροπίες, κουλτούρες και είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μία μοναδική ε, πολιτική κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Σύντομη. Εγώ λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί μια τόσο φιλόδοξη ε, πρόταση πρωτοβουλίας ε, ε, κατέληξε με αυτόν τον τρόπο που κατέληξε. Και θεωρώ ότι κατέληξε εκεί που κατέληξε για λόγους που υπόθηκαν από τους συναδέλφους ότι η ιστορία πρέπει να παραμένει ανεξάρτητη για τους ιστορικούς ε, αλλά και από την πολύ φανερή προσπάθεια του εισηγητή να περάσει μια εμπειρία ε, σε ε, ένα κοινό, σε άλλους συναδέλφους που όχι πως δεν αναγνωρίζουν αυτά που συνέβηκαν εκεί αλλά που θα μπορούσε νομίζω να τα δει με μια υπέρβαση όπως η γενιά της ε, γερμανικής κοινωνίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετώπισε το ναζιστικό τους παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν ότι αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να γράψουμε την ιστορία. Καλά είναι να την αφήσουμε στους ιστορικούς. Αλλά αν θέλουμε να κρατήσουμε τη συνοχή σε αυτό το κοινοβούλιο που αντανακλά τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας και να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το παρελθόν όχι προκειμένου να κατοχυρώσουμε τη δική μας ιστορική άποψη αλλά για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα. Τελευταία ομιλήτρια, η συνάδελφος Τρουπελ. Μόνο μία παρατήρηση, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν ε, σημαντικοί λόγοι για να καταδικάσουμε τα εγκλήματα του σταλινισμού και του κομμουνισμού. Ξέρουμε τι τρομερές ε, θηριωδίες και εγκλήματα έγιναν στα Γκουλά και τα στρατόπεδα συγκέντρωση. αλλά με βάση αυτά τα οποία αποκαλούμε στη Γερμανία η διαμάχη των ιστορικών, υπάρχει υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι, τα εγκλήματα του ναζισμού, του εθνικού σοσιαλισμού και την προσπάθεια εξολόθρευσης λαών και κοινοτήτων να τα θεωρούμε ως την απόλυτη έκφραση του, ε, απολυταρχισμού και να μην τα θεωρούμε ισότιμα με τα εγκλήματα του σταλινισμού. Αυτό θα ήθελα να ε, ε, το λέει η έκθεση και αυτό ήταν μια ε, επίκρισή μου. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Να κλείσω τώρα τη συζήτηση που νομίζω πως έγινε πολύ σοβαρά. Ίσως θα έπρεπε να γίνει προηγουμένως. Ευχαριστώ όλους που ε, συμμετείχαν και από κανέναν δεν αφαιρώ το δικαίωμα ε, να λέει ότι αντιμετώπισε σοβαρά το θέμα αυτό. Θα είχα προτιμήσει να είχαμε καταλήξει σε μια έκθεση που να μας είχε βοηθήσει όλους λίγο περισσότερο. Αλλά ό,τι έγινε έγινε, ίσως στο μέλλον να τα πάμε καλύτερα. Δεν αντιμετωπίσαμε αυτή την έκθεση ως ιστορική, την αντιμετωπίσαμε ως πολιτική από διάφορα έθνη, από διάφορες, ε, με διάφορες παραδόσεις, με, διάφορες, με διαφορετικές παραδόσεις, με διαφορετικές εμπειρίες και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο τελικά να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που να μας ενώνει όλους. Ήταν αμφίροπη η πλειοψηφία, η, το αποτέλεσμα ε, για λίγους λόγους απερίφθη, αλλά Νομίζω ότι αυτό έγινε επειδή όλοι θα ήθελαν να έχουν περιληφθεί άλλα σημεία στην έκθεση. Ευχαριστώ όλους που με καλή θέληση συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και κλείνω αυτή τη ε, συζήτηση τώρα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Έχετε τις αποφάσεις των συντονιστών. Αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν υπάρχουν ε, άλλα σημεία. Στις 25 Ιανουαρίου έχουμε την επόμενη συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου. Ε, συγγνώμη, 20 και 21 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Εύχομαι σε όλους ειρηνικά Χριστούγεννα και ε, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay.